Πάμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Έκθεση Φέρμπερ. Η αγορά χρηματοστατικών μέσων. Συνάδελφε Πόλτσακ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ υποστήριξα την έκθεση γιατί αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ναι, πρόεδρε, σας παρακαλώ όμως, ε, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τόση φασαρία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω λοιπόν να πω πως ε, ε, ενέκρινα τις δύο εκθέσεις του κυρίου Φέρμπερ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθεί να παρακολουθεί και να καθιστά λειτουργική την εσωτερική αγορά ακόμα και αν τα νέα κράτη υψώνουν νέους φραγμούς είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει την αναθεώρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων στις ε, εμπορικές αγορές. Σας ευχαριστώ. Ε, la parola sempre a lei, onorevole Polciak, prego, anche qui per un minuto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 είναι για να εξασφαλιστεί, για η ασφάλεια δικαίου. Είναι απαραίτητο τελικά να δοθεί αυτή η παράταση για να αντιμετωπίσουμε τις ε, καταχρήσεις στην αγορά. Ευχαριστώ. Αλλά όχι τελικά ε, για την έκθεση Χόιμπουχ ο κύριος Μαούλου. Παρακαλώ. Πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση αυτό το διάταγμα. Θέλουμε μια συμμαχία για μια βιώσιμη γεωργία, συμμαχία για τα τρόφιμα και θα πρέπει να είναι ένα στόχο αυτή τη Ευρώπη που έχει διάφορα τυπικά προϊόντα, κυρίως στον τομέα αυτών που σήμερα παρουσιάσαμε είναι και ισχυρό σημείο, πάρα πολύ ισχυρό σημείο της Ευρώπης αυτός ο τομέας. Ευχαριστώ συνάδελφε Μαγκίνες, έχετε το λόγο και εσείς για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υποστήριξα την έκθεση ιδιαίτερα εκεί όπου ζητεί από τις χώρες να θεσπίσουν δεσμευτικά νομοθετήματα για την υφαρπαγή γεώνα και πιστεύω ότι πρέπει και στο θεματολόγιο για την αναπτυξιακή πολιτική, για τα τρόφιμα, για τη διατροφή να καλύψουμε και θέματα γεωργικών γεών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν την επιλογή για το τι θα χρησιμοποιούν ως μέσον ανάπτυξη τεχνολογία. Αυτό το είδος, η επιλογή μιας τεχνολογικής εξέλιξης είναι δικαίωμά τους. Σε αυτές τα τεχνολογικά μέσα περιλαμβάνεται και η ε, τηλεκαταγραφή γεών για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ Μακοβέ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μια μεγάλη οργάνωση, η ένα, ένα FSN που χρηματοδοτείται από την G8 επιδιώκει να ε, υποδουλώσει τα φτωχά αφρικανικά κράτη. Εμείς θέλουμε να τα βοηθήσουμε για να σταματήσουν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Θέλουμε να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και να μπορέσουν ε, τα αφρικανικά κράτη να παράγουν και να διαθέτουν τα γεωργικά τους προϊόντα σωστές τιμές. Παρακαλώ λοιπόν και καλό τους ηγέτες του G8 να μην υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες για εφαρπαγή των γεών. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη γεωργία και την δίκαιη κατανομή των πόρων στα κράτη αυτά. Ο κύριος Κέλλη έχει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ Εργάστηκα ως θελοντή στο Μαλάουι πριν από μερικά χρόνια και ξέρω πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Καταλωσούριζω λοιπόν την έκθεση. Και θα την υπερψηφίσω, ελπίζω όλο το ΕΛΚ να το πράξει. Πρέπει να υποστηριχθεί η γεωργική οικονομία, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και οι πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τους όρους διαβίωσης των οικογενειών των γεωργών στην υποσχαχάρια Αφρική. Πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μικρές οικογενειακές ιωρικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις. Πρέπει να προαχθούν συστήματα ηλεκτρονικής τεχνολογίας που θα βοηθήσουν και στην καλύτερη διαχείριση των γεών, η παραγωγή και βέβαια θα αντιμετωπίσουν τη χρόνια, τους χρόνιους λοιμούς στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Στόλογιαν η έκθεση με την κυρία Μακοβέη. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Η παραποίηση λογιστικών βιβλίων ε, των επιχειρήσεων θέτει σε κίνδυνο την οικονομία ολόκληρη ενός κράτους. Γι' αυτό χρειάζονται ίδια πρότυπα λογιστικά σε όλες τις χώρες. Θέλουμε σαφείς, ξεκάθαρους δρόμους για την καταγραφή των ε, δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών. Υπάρχουν άλλωστε τα πρότυπα αυτά. Έχει γίνει πολλή δουλειά σε σχέση με τα διεθνή επιχειρηματικά, ε, λογιστικά πρότυπα. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με 14% ως μεγαλύτερος χορηγός στο σχετικό Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει λοιπόν και να αναθεωρούνται ή να επανεξετάζονται τα λογιστικά πρότυπα όσο το δυνατόν ε, ε, σε αιτήσια βάση. Ευχαριστώ Βαν και έχει το λόγο ο κύριος Πόψιλ που δεν είναι εδώ όμως οπότε παρακαλώ την κυρία Μακοδέη ένα λεπτό να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, η ανάδειξη τρομοκρατικών ομάδων στη Σομαλία, την Ιγυρία, στην περιοχή του Σαχέλ έχει ανατρέψει το κλίμα το σχετικό με την ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Τρία δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του χρηματοπιστωτικού μέσου για την ειρήνη στην Αφρική συμβάλλουν τα κράτη της Ένωσης. Είναι ως εκ τούτου ο μεγαλύτερος χορηγός για τις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. Ωστόσο, οι αποστολές αυτές δεν χαρακτηρίζονται από συνθήκες διαφάνειας. Δεν ξέρουμε τι γίνονται τα χρήματα αυτά. Τα μέσα, λοιπόν, για τη διαφύλαξη, για τη διατήρηση της ειρήνης, η χρηματοδότηση αυτή, δεν ξέρουμε ούτε εάν θα είναι, αν θα μπορεί να διατηρηθεί σε αηφόρο βάση, ούτε πώς διατίθεται. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, λοιπόν. Διαφάνεια στην καταγραφή των ποσών και των δαπανών, και πρέπει τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την ασφάλεια στα αφρικανικά κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μπόρεσα να υποστηρίξω αυτή την έκθεση μαζί με την ομάδα μου. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην ε, Αφρική, Υποστηρίζεται την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ. Εστιαζόμεθα στη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Λέμε ότι εγγυητή τη ειρήνη και ασφάλεια είναι ο ΙΕ σε διεθνέ επίπεδο. Πάνω από 120.000 άτομα είναι σε όλο τον κόσμο μέλη του ΙΕ. Οι περισσότεροι από αυτού υπηρετούν στην ε, Αφρική σε ειρηνευτικέ αποστολέ. Ο βασικό μηχανισμό συνεργασία με την Αφρική είναι το μέσο ειρηνή στην Αφρική. Το πρόγραμμα δράση καλύπτει τα διάφορα κενά που έχει αυτό το μέσο και δείχνει διαφόρου διεξόδου και επιμερισμό των, ε, του βάρου με τα χώρε Αφρική ε, διευκόλυνση διαδικασία λήψη αποφάσεων και στοχευμένε δράση. Θέλουμε αυτό το μέσο να είναι είσοδο για τη δημιουργία ισχυρότερη ε, σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Αφρικανικής Ενώσεω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Έκθεση Τσέζακ. Συνάδελφε Μαγκίνες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ λακωνική και να πω ότι εκ μέρου τη Επιτροπή Γεωργία καλωσορίζουμε την υποστήριξη που δέχτηκε αυτή η έκθεση. Συνεργαστήκαμε με του συναδέλφου του ΣΥΜΚΟ και τονίζει σαφέστατα ότι πάνω από 600 μέλη του Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερε δράσει για να αντιμετωπίσουμε τι εμπορικέ πρακτικέ στον τομέα των τροφίμων. Στέλνουμε έτσι ισχυρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλου του ενδιαφερόμενου φορεί ε, τη ασία τροφίμων για τι πολιτικέ ανησυχίε που έχουμε όσον αφορά το θέμα αυτό. Κανεί από εμά δεν έχει την ιδεώδη λύση. Όλοι μα έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα που υφίστανται και όπου υπάρχει ανισορροπία εξουσία στι δύο άκρε αλυσίδα τροφίμων. Αυτή η έκθεση, όπω σα είπα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα ε, ακούσει αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ συνάδελφε Μαγκίνας, συνάδελφε Μαούλου. Έχετε ζητήσει το λόγο, δεν είναι στην αίθουσα όμω. Συνάδελφε Λόπες Μπερμέιο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απέσχουν όσον αφορά αυτή την ε, έκθεση για τι αρέντες πρακτικές όσον αφορά τα αγροδιατροφικά θα πρέπει να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους και τους ε, γεωργού όσον αφορά τη χειραγώγηση των ε, τιμών όσον αφορά ε, την διανομή των προϊόντων γιατί είναι πάρα πολύ ευάλωτε, πάρα, πολύ μετάβολες τιμέ σε αυτή την αλυσίδα και αυτό είναι αλυσίδα δηλαδή διανομής και αυτό είναι μεγάλη απειλή οπότε έχουμε αυτές τις αλυσίδες της διανομής που κινείται μέσα στα πλαίσια της ε, ΚΑΠ, αλλά τώρα έχει γίνει πιο έντονη ο ανταγωνισμός μεταξύ των γεωργών, γιατί έχει γίνει απορρίθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, διεθνείς συναλλαγές. Όλα αυτά έχουν γίνει επίτηδες και έτσι έχει μόνιμο χαρακτήρα η αστάθεια των γεωργικών αγορών και έτσι επίσης υπάρχει διαρθρωτική έλλειψη ισορροπίας και ανισότητα μεταξύ των μεγάλων ε, ε, μονάδων διανομής και των ε, ε, γεωργών. Έτσι έχουμε απορρίθμιση του εμπορίου. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κάπου που να έχει ως επίκεντρο την παραγωγή και τώρα που υπάρχει κρίση στις τιμές αυτή κάπου να δίνει λύσεις. Νέκοφ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές εμποδίσουν την ανάπτυξη της παραγωγής και, της, ιδιαίτερα της παραγωγής τροφίμων. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και ακριβώ τα προβλήματα αυτά οδηγούν στην ε, αποδιάρθρωση και ουσιαστικά καταστροφή ενός ολόκληρου τομέα. Αυτές οι αθέμητες πρακτικές προξενούν τεράστιες ζημιές στους γεωργούς και τελικά καταλήγουν στην ε, πτώχευση πολλές εκμεταλλεύσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν η παραγωγοί να έχουν συνθήκες θεμητές αγορέ, αγοράς, δηλαδή να εξασφαλίζουν και τις τιμές αγοράς ως ε, αμοιβή για τα προϊόντα τους για να μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους και να έχουμε έτσι καλύτερη αγορά προϊόντων στην ε, Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την έκδοση αυτή, με την εκδοχή αυτή του κειμένου. Νομίζω ότι Πρέπει να σταματήσουν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Γιατί γίνονται πολλές χειραγωγήσεις των αγορών όπου οι μεγαλύτεροι έμποροι, χονδρέμποροι μπορεί να καταστήσουν πολύ δύσκολο το έργο και την επιβίωση ακόμη των μικρότερων. Εδώ οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, ε, το λιανεμπόριο είναι ε, αρτηρία ζωτική για την αγορά των τροφίμων και πρέπει να μην τις αφήσουμε στη μοίρα τους. Πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά και εδώ έχουμε να κάνουμε μια από τις κυριότερες αρχές, δηλαδή την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του καταναλωτή με όρους διαφανής σε σχέση με, την, ε, με τις ε, πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφιμών. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο, παρακαλώ. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί. Μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 εξηγεί ότι αυτές οι πρακτικές υφίσταται σε όλα τα μέρη της αλυσίδας ε, των τροφίμων. Υπάρχει ανισορροπία μεταξύ ε, των διαφόρων φορέων και τη θέση εξουσία. Ε, και αυτό είναι ει βάρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μικρή παραγωγή όμως αποτελούν περίπου το 90% της οικονομικής δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι πιο ευάλωτοι αυτοί που έχουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σίγουρα ε, είναι δύσκολο να επιβιώσουν στην αγορά, κυρίω λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που υπάρχει. Είναι Μπορούν να προταθούν μάλλον καινούριε πρωτοβουλίες. Ε, ε, χρειάζεται μια αγορά που να είναι πραγματικά ελεύθερη και γι' αυτό η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ανταγωνισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ούτω ώστε να μπορεί να αντιταχθεί στον αθέμητο ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μαζί με την ομάδα μου ψήφισα στις τρεις ψηφοφορίες αυτή την έκθεση η οποία θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές αθέμητες αυτή η λέξη αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά τι πρακτικέ που ακολουθούνται, ποιε είναι οι λύσει ώστε να δώσουμε στου γενοπολιτέ και στου παραγωγού τροφίμων προστασία κατά των αθέμητων εμπορικών αυτών πρακτικών. Εξετάσαμε θέματα όπω αποτελεσματικότητα θελοντικών σχημάτων ε, τι γίνεται με την παραγωγή με ιδιωτικών προϊόντων ε, και τέθη μεγάλο ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένη προσέγγιση νομοθετική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όχι. Τελικά η Επιτροπή και το ΕΛΚ αποφάσισαν, αποφασίσαν ότι θέλουμε θελοντικά σχήματα εντοπίζοντας πρακτικές αθέμητες αντιμετωπίζοντα όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ελπίζουμε ότι η έκθεση θα οδηγήσει σε εξάλληψη των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, αλλά θα... Ε, περιμένω. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, περνάμε στην έκθεση Μάκιντάερ. Ο συνάδελφος Μαουλού που έχει ζητήσει το λόγο δεν είναι παρόν. Πάμε στην κυρία Μαγκίνες. Έχετε το λόγο, κυρία Μαγκίνες. Ναι, συμπαθάτε με κύριε Πρόεδρε. Έχω το λόγο. Α, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, μιλήστε. Θέλω να επισύρω την προσοχή σε σχέση με αυτή στην παράγραφο 74. Εκεί μνημόνεται η ανάλυση με τη βάση του κινδύνου και τη μερόληπτη ε, ανάλυση αυτού. Οπότε κοιτάξτε να δείτε ποιοι, τι λέει η ανάλυση κινδύνου και τι πρέπει να γίνεται σχετικά. Αλλά επίση θέλω οι συνάδελφοι να ρίξουν μια ματιά και στην παράγραφο 33. Λέμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι γεωργοί ε, μπορούν να είναι ενημερωμένοι για αυτές τις ε, τεχνικές και να υπάρξει επίσης δημοσία συζήτηση για τα εν λόγω ζητήματα. Άρα θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε αυτό να πραγματοποιηθεί γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε ενημέρωση του κόσμου σε σχέση με τις τεχνολογικές ε, λύσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές υπήρχε αντίσταση ε, κατά αυτών των ε, λύσεων. Να μην ξαναγίνει αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μαγκίνες, λέει ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Νιάκοφ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ δεν υποστήριξα την έκθεση αυτή γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κενό δικαίου και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πρέπει να ε, σταματήσει αυτή η ασάφεια, πρέπει να μην στέλνουμε εσφαλμένα μηνύματα στον καταναλωτή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε τέτοια περιθώρια ε, ανα, αμφιβολία σε σχέση με την εισαγωγή ή μη ε, τέτοιων πρακτικών. Ο τομέας αυτός της γεωργίας μας αφορά όλους. Έχουν να κάνουν με, έχει να κάνει με τα τρόφιμα, με τα φυτά τα οποία θα καταναλώσουμε ως τρόφιμα και έτσι δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, τέτοιες ελλείψεις. Πρέπει να βρούμε λύσεις αποτελεσματικές για τον καταναλωτή, για τους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Νικέλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ζήτηση για τρόφιμα ε, αναπτύσσεται και φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί μέχρι το 2070 κατά 20%. Δηλαδή είναι τεράστιες οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει η γεωργία παγκοσμίω και πρέπει να παράγει περισσότερα τρόφιμα και πρέπει να περιορίσει τις ανάγκες αιγαίες και πρέπει να αντιμετωπίσει λειψιδρίες, ε, κινδύνους που προκύπτουν από νέα, νέα ζυζάνια, νέα νέους παράγοντες ζημιογόνους για τη φυτική παραγωγή και το καθεξής. Άρα περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη αηφορία θα χρειαστούν για να μπορέσει ο γεωργικός τομέας να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αυτές προκλήσεις. Έχουμε ένα παλόμενο γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τεχνολογίες, οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε κάθε τύπο γεωργικής παραγωγής. Οι, οι, Ιρλανδικές επιχειρήσεις είναι στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας χρόνια τώρα και υποστηρίζουν έτσι έναν ισχυρό Ιρλανδικό γεωργικό τομέα που αξιοποιεί τόσο πολύ καλά τις νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέλλη, λέει ο Πρόεδρος. Έκθεση Χόιτομα. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μαουλού. Πάμε στην κυρία Τόρες Μαρτίνες. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν απειλείται γιατί δεν έχει καινοτομία. Απειλείται από αυτές τις συνθήκες ελευθερών εμπορίου που κλείνονται εγκρυπτό και παραβίστο πίσω από τις πλάτες του κόσμου και στην ε, Ισπανία. Έχουμε υψηλή τεχνολογία. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει και καταστρέφονται οι γεωργοί βέβαια και χρειάζεται η καινοτομία για να δημιουργηθεί ευμάρια και πλούτος και βέβαια θα πρέπει η Ευρώπη να δημιουργεί συνθήκες ούτως ώστε η ύπεθρος να ε, έχει καινοτομία όμως αυτό είναι και ένας ε, μύθος όσον αφορά αυτές τις ε, συνθήκες τις συμφωνίες θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ρίζα του κακού για την Γεωργία είναι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε το μοντέλο, το πρώτο παραγωγής που έχουμε γιατί δίνονται χρήματα σε προγράμματα τα οποία ε, καταρρύπτουν την ε, αυτάρκεια της παραγωγής. Μόνο αν στηρίξουμε τους παραγωγούς θα έχουν αυτοί μέλλον και θα έχει μέλλον και η ύπεθρος. Κύριε Νιέκοφ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Προστήριξα την έκθεση διότι είμαι πεπισμένος πως η αηφόρος αξιοποίηση των πόρων της γεωργίας έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει και η τεχνολογία για τη βελτίωση της παραγωγής της γεωργίας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από τα παραδοσιακά λοιπάσματα και να ενισχύσουμε έτσι τη βιολογική γεωργική παραγωγή για να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και τα εδάφη της ε, γεωργίας. Καλό λοιπόν όλους τους βουλγαρούς συναδέλφους να υποστηρίξουν τις προτάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν και να προστατεύσουμε τη Μαύρη Θάλασσα. Μια λύση καλή για επενδύσεις, καλύτερες για καλύτερη γεωργία, για καλύτερες για οικονομικές δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Κόρατσα λεπτό. Το Πρόεδρε, ζητάμε εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας σαν Ευρωκοινοβούλιο. Είναι καλύτερο τρόπο να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές. Επίσης, καλωσορίζω το ότι θα ξαναθέσουμε σαν θέμα και την σπατάλη των τροφίμων. Αποτελεσματική γεωργία είναι σημαντική για να θρέψουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό του κόσμου. Είναι εξίσου σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα παραγόμενα. 100 εκατομμύρια τόνοι φαγητού χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο και αυτή η σπατάλη των τροφίμων είναι κάτι απαράδεκτο και ηθικά και οικονομικά. Λοιπόν, το τονίσαμε αυτό και θα πρέπει να αυξήσουμε τις δράσεις μας ε, επί δεκαετίε, Πρέπει να ηγηθούμε, να διαμορφώσουμε την κοινή γνώμη, να συνεργαστούμε με όλα τα μέρη της τροφή μα, του παραγωγού, του λιανοπολιτέ και του καταναλωτέ. Όλοι πρέπει να υπομισθούμε τι ευθύνε μα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μα και τη στάση μας του φαγητού σε επίπεδο προκυσενό. Χρειαζόμαστε κοινού ορισμού, καλύτερη συλλογή στοιχείων, στόχου, ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διευκρίνηση ημεριομηνιών λήξεω στι ετικέτε. Και θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιεί το και ε, για βοήθεια Λοιπόν, είναι κοινή πρόκληση το πρόβλημα αυτό των τροφίμων. Δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι μια επιλογή αυτή που ακολουθούμε, αλλά ότι είναι μια αναγκαιότητα να αλλάξουμε. Ευχαριστώ, Άννα Μαρία. Συνάδελφε Κέλλη, τελευταία παρέμβαση. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα πρόβλημα να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση, λέει ο κύριος Κέλλη, και πραγματικά μοιάζει πολύ με την προηγούμενη έκθεση για τη γεωργία. Λοιπόν, θέλουμε βιώσιμη γεωργία. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές προοπτικές των παραγωγών. Πρέπει η οικονομική ανάπτυξη, η βιώσιμη παραγωγή να μην αποκλίνουν το ένα το άλλο. Χρειάζεται καινοτομία και έρευνα. Σημαντικό ρόλο του για την επίτευξη των στόχων. Θέλουμε καλύτερε προοπτικέ οικονομικέ και βιώσιμη παραγωγή. Μικρομεσαίε εκμεταλλεύσει. Τεράστια σημασία παίζουν στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Πρέπει λοιπόν τα ωφέλη τη καινοτομία και τη έρευνα στη Γεωργία να φτάνουν στι μικρομεσαίε εκμεταλλεύσει δεν πρέπει να ωφελούνται μόνο οι μονάδε μεγάλη παραγωγή. και θα πρέπει και οι ορεινέ περιφερειακέ περιοχέ να προστατευτούν. Αυτέ που είναι σε δυσχερή θέση θα πρέπει να ωφεληθούν έρευνα και τενοτομία. Σημαντική γεωργία για τη χώρα μου. 9 δι εξαγωγέ, 10% των εξαγωγών ε, και για πάρα πολλέ οικογένειε που εργάζονται στον τομέα τη γεωργία και θρέφονται. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση ήταν η δική σα, κύριε Κέλλη. Δεν απομένει παρανακοινώσω ότι διακόπτεται η σύνοδος μέχρι τις 3. Γεια σας.